την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία. Ελπίζω να με βοηθήσετε να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να σας ξαναδώ στην επόμενη μέρα του 2012. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της εκθέσεως ΣΒΕΡ ε, νεολαία σε κίνηση. Εγώ την θέτω σε ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προβλέπετε τώρα ψηφοφορία της, του ψηφίσματος της κυρίας Χάνιμπολ τη θέτω σε ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλες και όλοι παρακαλώ πέρας εγκρίνεται και συγχαίρω και τους δύο εισηγητές για την έκθεσή τους. Προβλέπεται τώρα ψηφοφορία πέντε προτάσεων ψηφισμάτων για την έγκριση του πρωτοκόλου για τη συνέχιση της ε, Συμφωνίας Ελίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Μαυριτανίας. Πρώτα δεν έχει υποβληθεί τροπολογία. Θέτω υπό σε ψηφοφορία λοιπόν την κοινή αυτή η πρόταση ψηφίσματο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και συγχαίρω την εισηγήτρια. Ψηφοφορία δύο προτάσεων ψηφισμάτων για ίση πρόσβαση στις αγορές δημοσίων προμηθειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρώ στην ψηφοφορία των ψηφισμάτων τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλά, θέλετε επαλήθευση λοιπόν. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 2. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία την πρώτη ψηφίσματο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφοφορία 7 προτάσεων ψηφισμάτων σχετικά με την κρίση στον ευρωπαϊκό τομέα αλληλείας λόγω της αυξήσεως των τιμών του πετρελαίου. Κοινή πρόταση ψηφίσματος 5 πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 2 Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. απερίφθη. Τρία. Νομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος τέσσερα. Ψήφι υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην πρόταση ψηφίσματος 6 πολιτικών ομάδων για το πρόγραμμα Small Business Act. Παράγραφος 9. Ε, χωριστή ψηφοφορία μάλλον, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 21 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29. Παράγραφος 29. Ψήφι υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Προφορική τροπολογία της κυρίας Τζαβέλα. Επιθυμείτε να θέσετε το προφορική τροπολογία κυρία Τζαβέλα. Η κυρία Τζαβέλα. Για συμβασμό σε μια κοινή τροπολογία που θα έχει ως εξής λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη παράνομη εμπορία σε όλες τις χώρες μέλη παραχαραγμένων ή πειρατικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και τα οποία απειλούν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όλοι οι συγγραφείς συμφωνήσαμε επί του κειμένου αυτού. Μάλιστα, υπάρχουν ενστάσεις. Εγερθείτε εάν έχετε ενστάσεις. Δεν βλέπω, άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 9 με την προφορική της κυρία Τζαβέλα. Ψήφι πέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το κοινό ψήφισμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ε, ψηφοφορία της εκθέσεως της κυρίας Μέρκιες Προηγουμένω, να συγχαρώ όλου ε, του συντάκτε του ψηφίσματο. Έκθεση σε Ένωση Καινοτομία μεταμορφώνεται στην Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση. Η κυρία Τσικάου θέλει το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα να ζητήσω από του συναδέλφου να υπερψηφίσουν την τροπολογία υπαριθμών 1 ναι, θα ήθελα να στήσω του αδέλφου να υπερψηφίσουν την τροπολογία υπαριθμών 1, διότι θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για την ε, πολιτική κοινοτομία Να διαγράψουμε όμω το funds from common agricultural policy. Ε, δεν υπάρχει συζήτηση, κυρία μου, τώρα. Συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια πρόταση. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία τη έκθεση Μέρκη. Με το σχέδιο ψηφίσματο. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Mm. Παράγραφος 128 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο στροποποιήθηκε. Ή μάλλον να κάνουμε μία επαλήθευση για την δεύτερη παράγραφο της 128. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος ε, για τη σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας με σύσταση σχετικά με τους υγειακούς βοηθούς. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τρία υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο ε, του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Γεωργίας για την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Περνάμε στην ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος, για την οποία δεν υπάρχουν τροπολογίες. Παράγραφος 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη R, υπέρ. Όχι, να κάνουμε μια παλήθευση για την παράγραφο 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη R υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση ΣΑΚΕΝ, πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ψηφίζουμε την παράγραφο 9 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 29 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 38 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Mm. Εγκρίνεται παράγραφος 50 σε δύο τμήματα και με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Σάκε. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Σάντσε Σμιθ, απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Περνάμε στην εξέταση. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Παράγραφος 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι και όλες. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το σύνολο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Σάντσε Σμιθ. Τελική ψηφοφορία, τελευταία για σήμερα δηλαδή. Το ψήφισμα για το Σαράγεβο ως πολιτιστική πρωτεύουσα το 2014. Δεν υπάρχουν τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Έληξαν οι ψηφοφορίες.